Bien, empezamos. Empezamos con la comisión eh, de peticiones y voy a darles. Κοινάει η συνεδρίασή μα. Έχουμε το πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις ε, από την συνεδρίαση των συντονιστών. Έλαβαν τις εξής αποφάσεις λοιπόν οι συντονιστές. Η ημερήσια διάταξη για τον Απρίλιο εγκρίθηκε με τις εξής αλλαγές. Ε, η 760 και η 323 ε, αναβλήθηκαν για τον Μάιο γιατί αναμένουμε εντωμεταξύ τις απαντήσεις από τις εθνικές αρχές και δύο γνωμοδοτήσεις. Μία για τις ε, διασυνοριακές ε, υιοθεσίε και μία, της Γιούρη και μία της Λίβη για την κατάσταση στην ε, Μεσόγειο. Θα μας απασχολήσουν μία ακρόαση στο δεύτερο εξάμεινο και θα γίνει άλλη μία ακρόαση μετά το πρώτο εξάμεινο του 2016 για τα θεμελιώδη δικαιώματα. και θα έχουμε και κρόση τον Ιούνιο μετά για το δικαίωμα στην αναφορά για τα δικαιώματα των παιδιών. Για την πρόταση του ΙΦΤΤ θα έχουμε ένα σεμινάριο ή ένα εργαστήριο αναλόγως για τις διαρνητικές αποστολές του 2015 θα σας ζητήσουμε να υποβάλλετε προτάσεις πριν από τις 10 Απριλίου όλες οι συστάσεις ε, που έγιναν από την ε, γραμματεία εγκρίθηκαν. Μετά υπάρχει το θέμα της Ιρλανδίας που έκλεισε, ζητήθηκε να ξανανοίξει, απορρίφθηκε. Μετά υπήρχε το πόρταλ, η πύλη διαδικτυακή, ζητήσαμε αντιδράσεις μέχρι τον Απρίλιο. Αυτές ήταν ουσιαστικά οι αποφάσεις της ε, συνεδρίασης ε, των συντονιστών και περνάμε τώρα στην ε, υπόλοιπη μερική διάταξη. Ναι, ο Μαριάς. Θα ήθελα και στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας να διαμαρτυρηθώ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η πρόταση του ECR για την διενέργεια δημόσιας ακρόασης για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις. Ήδη σε προηγούμενη συνεδρίαση το αίτημά μας για την διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης καταψηφίστηκε από τον συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την συντονίστρια του S&D. Ψηφίστηκε το αίτημά μας εκείνο από τους συντονιστές του ECR, δηλαδή εμένα, την πρόταση που έκανα, του EFD και της ΓΚΟΕ. Και οι δύο υπόλοιποι συνάδελφοι έκαναν αποχή. Σήμερα λοιπόν που ξανατέθηκε το ζήτημα σε συζήτηση και ψηφοφορία, αυτό που έγινε και για το οποίο διαμαρτυρήθηκα και διαμαρτύρομαι και εδώ, είναι ότι δεν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρότασή μας. Με ένα διαδικαστικό τρίκ διαμορφώσατε εσείς ως πρόεδρος μία πρόταση πακέτο για το ποιες δημόσιες ακροάσεις θα γίνουν το δεύτερο εξάμεινο του 2015 και αρχές του 2016 και την δική μας πρόταση δεν τη συμπεριλάβατε σε αυτό το πακέτο, την απορρίψατε και ζητήσατε να γίνει ψηφοφορία επί της προτάσεως πακέτο. Σε αυτήν την ψηφοφορία απήχα, διότι δεν ήθελα να νομιμοποιήσω τις ενέργειες του Προεδρείου, η οποία ενέργεια του Προεδρείου δεν έθεσε σε ψηφοφορία την πρότασή μας προκειμένου να πάρουν την ευθύνη όσες πολιτικές ομάδες πιστεύουν ότι ήθελαν να καταψηφίσουν την πρόταση για δημόσια ακρόαση για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ήταν ένα διαδικαστικό τρίκ, το οποίο όμως στέρισε το δικαίωμα σε εμά να έχουμε μία ψηφοφορία επί της προτάσεώς μας. Γι' αυτό λοιπόν διαμαρτύρομαι, επισημαίνω ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι το θέμα, θα ασκήσουμε κάθε πολιτικό και νομικό μας δικαίωμα, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όποιες πολιτικές ομάδες θέλουν να καταψηφίσουν την πρόταση για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις πρέπει να έχουν το θάρρος να το κάνουν κανονικά και όχι να κρύβονται πίσω από διαδικασίες και τρίκ ούτω ώστε να αποφεύγουν να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν όπως ήθελαν την πρότασή μας. Ξέρουμε ότι οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στην Ευρωβουλή, του Σοσιαλιστικής Ομάδας στην Ευρωβουλή, έβγαλαν ανακοίνωση, ενώ δεν όφυλαν και δεν τους κάλεσε κανείς, με την οποία έπαιρναν θέση υπέρ της Γερμανίας και κατά της Ελλάδος στο θέμα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων όταν τέθηκε επίσημα την ελληνική κυβέρνηση πριν λίγο καιρό. Ας έχουν λοιπόν το θάρρος να το τοποθετήσουν και εδώ. Γι' αυτό παίρνω αυτή τη θέση, εξηγώ ότι διαφωνώ με τις αποφάσεις των συντονιστών και δημοσίως θέτω το θέμα αυτό στην Επιτροπή, επιφυλασσόμενος για το τι ενέργειες επί του θέματος αυτού θα κάνουμε ο ECR και πολιτικά και νομικά. Ευχαριστώ. Bueno, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πως ε, αισθάνομαι ε, κάπως να απειλούμε και ειλικρινά αυτά τα οποία λέτε δεν ισχύουν. Δεν είναι ε, γεγονός πως θέλω οι σοσιαλιστές ε, να κατονομάζονται σε αποφάσεις σε οποίες δεν συμμετείχαν. Εγώ εξήγησα την ε, ψήφο μου, την αιτιολόγησα, εξήγησα γιατί ψήφισα το πως ψήφισα και είπα πως ναι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα, αντι, αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία αυτή, αλλά συνεχίζετε να το ε, φέρνετε και συνεχώς λέτε τα ίδια πράγματα. Εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε, αλλά το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα ήδη στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να ζητήσω από την Πρόεδρο να μην ξανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πέτερ. Ήθελα να συμπληρώσω μόνο το εξή. Έχουμε ένα σημείο ε, στο σημείο 6 τώρα. Κοιτάξτε, υπήρχαν διαφορετικές προτάσεις και είναι υποχρέωση της Προέδρου να καταλήξει, να συμβιβάσει κάποιες αυτές τις προτάσεις. Έγινε ένα πακέτο λοιπόν, έγινε μια ψηφοφορία πακέτο. Καλύπτεται αυτό από τον κανονισμό, το πακέτο αυτό ψηφίσαμε και δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως είπα δεν είναι δικαίωμα, αλλά υποχρέωση της ε, Προέδρου να καταλήγει σε ένα συμβιβασμό. έξι νομίζω τροπολογίες είχαν προταθεί και νομίζω πως ε, κατέληξε ένα καλό συμβασμό η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πίτερ, ο κύριος Μαριάς. Ανεξαρτήτως του ποια ήταν η αιτιολογία της συντονίστριας της σοσιαλιστικής ομάδας στην προηγούμενη ψηφοφορία μας, σημασία έχει ότι καταψήφισε την πρότασή μας. Δεν έχει σημασία τι λες, σημασία έχει τι ψηφίζει. Δεύτερον, αυτό που έθεσα σήμερα έχει σχέση με τα δικαιώματά μας ως βουλευτών και ως πολιτική ομάδας. Υποβάλαμε μία πρόταση και θέλαμε μία ψηφοφορία επί της προτάσεώς μας. Να ξέρουμε πολιτικά ποιοι ψηφίζουν κατά της δημόσιας ακρόασης για τις γερμανικές πολεμικές συμπανορθώσεις και ψηφίζουν υπέρ αλλά επειδή την προηγούμενη φορά εκτέθηκαν με την ψήφο τους κάποια πολιτικές ομάδες, το Λαϊκό Κόμμα και η Σοσιαλιστική Ομάδα, τώρα με την διαδικασία πακέτο ήθελαν να κρυφτούν. Σας λέω λοιπόν ότι πολιτικά δεν μπορείτε να κρυφτείτε για την αρνητική σας στάση και διαδικαστικά μας στερήσατε το δικαίωμα να έχουμε μια ψηφοφορία επί της προτάσεώς μας. Αυτό λοιπόν θέσαμε σήμερα, this time. Σήμερα θέσαμε το δικαίωμά μας να υπάρξει ψηφοφορία επί της νέας προτάσεώς μας. Αυτό δεν έγινε με το τρίκ περί προτάσεως πακέτου. Ευχαριστώ. Bien, doy por zajado este tema. La presidenta ha hecho el reunión de coordinadores. Λοιπόν, ε, η πρόεδρος ε, κατέθεσε μια πρόταση, υπέβαλε την πρόταση στους συντονιστές. Η πλειοψηφία των συντονιστών υπερψήφισαν την πρόταση, έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε και αληθεύει ότι ψηφίστηκε η πρόταση στην προηγούμενη σύσκεψη των συντονιστών, καταψηφίστηκε και σήμερα υπενθυμίσαμε την θέση σας στα πλαίσια της ψηφοφορίας για το πακέτο. Διαφωνούμε, ε, αποκλίνουν οι απόψεις μας, έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη των συντονιστών, πρέπει να προχωρήσουμε. Προτείνω να το σημείο 16 να το δούμε στις ε, 3 η ώρα. Παρακαλώ, κύριε Βαλέσσα. Το, ε, ζητώ τα σημεία 9 και 10 να συνδυαστούν, διότι είναι ίδιο το αντικείμενο και είναι λογικό να συζητήσουμε μαζί τα δύο σημεία. Ναι, ναι, αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι συντονιστές ε, θα συνδυάσουμε αυτά τα δύο σημεία και το 16 στις 3 θα το συζητήσουμε. Πολύ ωραία. Θα εγκρίνουμε τώρα τα πρακτικά. Τα έχετε όλοι λάβει. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 4. Οι ανακοινώσεις. Η πρωτοβουλία για την ε, ε, ηθαγένεια, την ευρωπαϊκή ηθαγένεια αποτέλεσε αντικείμενο συλλογής υπογραφών και άρα ε, εφόσον συγκεντρώθηκε ένα εκατομμύριο υπογραφές θα διοργανηθεί μια ακρόαση θα συνεργαστούμε με την, ε, τις Επιτροπές Άγκρη και Ήτρε βάσει του άρθρου 111 στις 11 Μαΐου του 2015 το απόγευμα θα δείξει αυτή η ακρόαση. Στείλαμε επίσης τον κατάλογο των μελών ό,τι έχει αποσυρθεί δηλαδή από τους αναφέροντες. Κρίνεται ότι υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, πέντε διάφορα δεν υπάρχουν, έξι ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών. Ε, έκανα την αναφορά των αποφάσεων των συντονιστών και φτάνουμε στο σημείο 7. Γνωμοδότηση σχετικά με την 30η και 31η τήση έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εγώ είμαι συγγήτρια. Θα βγάλω λοιπόν το καπέλο της Προέδρου για να σας μιλήσω για αυτή την έκθεση που υποβάλλουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ζητείτε ετησίως ε, μια τέτοια έκθεση από την Επιτροπή Αναφορών σε σχέση με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χαιρόμαστε που ε, το λένε και μεγαλύτερη σημασία στις αναφορές οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί παράβαση από πλευράς των κρατών μελών παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναφοράς από πλευράς των πολιτών στο τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας, της κατανάλωσης, της εσωτερικής αγοράς και ελεύθερη κυκλοφορία ε, των προσώπων ως επιτοπλίστων. 1.434 υποθέσεις ήταν ακόμη ανοιχτές. Όπως μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει μειωθεί όμως ο αριθμός των ανοιχτών υποθέσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο τα κράτη-μέλη συμμετέχουν ε, στο πιλωτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, που στόχο έχει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και χαιρόμαστε και για την προσήλωση αφοσίωση που δείχνουν οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή Αναφορών. Είμαστε υπέρ ε, επικοινωνιακής πολιτικής σε σχέση με τις αναφορές που ανοίγουν 30 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών. Δεν είχα χρόνο ακόμη για να συμπεριλάβω τις προτάσεις ε, των πρασίνων, ε, διότι περιμένω κάποιες μεταφράσεις. Σίγουρα θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο συμπεριλαμβάνοντας τροπολογία των και τον ΔΕΗ Δεν είμαι σκιώτης εισηγήτρια για αυτή την αναφορά η συνάδελφος η υπεύθυνη είναι λύπης αποστολή, αλλά έχω κάποια σχόλια. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σπέρα για τη δουλειά που έκανε, έξοχη δουλειά της, και για την επικοδομητική συνεισφορά της την ευχαριστώ. Πρέπει πράγματι να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Είμαι υπέρ των σχετικών μέτρων. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση. Η έκκληση αφορά την νομοθεσία και τις διαδικασίες τις σχετικές που ακολουθούνται. Εν γέννη, έχουμε 28 διαφορετικά νομικά συστήματα. Άρα για τους πολίτες είναι δύσκολο να γνωρίζουν που βρίσκονται όταν μετακινούνται από χώρα σε χώρα και κυρίως στον εμπορικό τομέα, στον επιχειρηματικό τομέα είναι πιο έντονο αυτό. Θα ήθελα να απευθύνω λοιπόν μια έκκληση ούτως ώστε η να γίνει η ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στι εθνικέ ενόμε τάξει. Θέματα υγεία, εσωτερική αγορά των υπηρεσιών, ε, οι διάφορε παραβιάσει είναι γνωστέ. Ε, και έχουμε αναφορέ σχετικέ με την μη συμπερίληψη, ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών στι εθνικέ ενόμε τάξει. Έχουμε θεσπίσει πολλούς νόμους, αλλά πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν τα δέοντα. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την εσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της εθνικές νομοθεσίας. Πρέπει ίσως να υπάρχει κάποιος άλλος μηχανισμός πέραν των κυρώσεων, να υπάρχει μια διαδικασία παρακολούθησης που θα επιτρέψει την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού ε, δικαίου στις εθνικές αναμεστάξεις, χωρίς να φτάνουμε αναγκαστικά στην επιβολή κυρώσεων. Συνοπτικά λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, θεωρώ ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ θετική και ότι η δουλειά είναι επικοδομητική. Υπάρχει άλλος συντονιστής που επιθυμεί να παρέμβει, λέει πρόεδρος. Όχι, αν δεν υπάρχει άλλος, θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ο Πέτερ. Äh, Πέρα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές γιατί είναι σημαντικό το θέμα και υποστηρίζω την πρόταση. Θα ήθελα να παρατηρήσω πως έχουμε πάντα το ίδιο πρόβλημα στην Επιτροπή Αναφορών γιατί πρέπει να συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν και έχουμε το πρόβλημα πως η επαφή, ο διάλογος ε, κομισιών και κρατών μελών δεν υπάρχει. Ανεφέραμε ένα παράδειγμα, έχω και άλλο παράδειγμα με την Τσεχία. Είχαμε θέσει ερώτημα από τον Οκτώβριο και δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα. Οπότε το ερώτημα προς την Κομισιόν είναι πώς θα βελτιωθεί αυτός ο διάλογος με τα κράτη-μέλη. Ποια είναι η εντύπωση της Κομισιόν. Τι είναι. Αρνούνται να συζητήσουν. Καθυστερούν. Τι κάνουν. Αν λοιπόν δεν λαμβάνουμε απαντήσεις ε, από τα κράτη-μέλη μέσω της Κομισιόν, δεν γίνεται τίποτα. Καρτάει πάρα πολύ η διαδικασία. Ξέρω πως δεν φταίει η Κομισιόν, αλλά κάπως θα πρέπει να παρακινήσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι. Θα υποβάλω και μία πρόταση για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πίτερ. Η Ιουλία για τους πράσινους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ πως η γνωμοδότηση πραγματικά αντικατοπτρίζει τη σημαντική θέση της Επιτροπής Αναφορών και το τι κάνουμε για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και χαιρόμαστε που ακούμε πως ε, κάποιες από τις προτάσεις ε, για τροπολογίες λαμβάνονται υπόψη και λαμβάνεται υπόψη και η εμπειρία που συγκεντρώνουμε στις περιπτώσεις αυτές και σημαντικό είναι η ε, Επιτροπή Αναφορών να εμπλέκεται από την αρχή στην ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω πως στις περιπτώσεις ε, παραβιάσεων όπου έχει υπάρξει κάποια απόφαση θα πρέπει η Κομισιόν να φροντίσει να εφαρμόζονται και στην πράξη αυτές οι αποφάσεις. Ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει η Κομισιόν. Ο κύριος Κέμπης, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να αντιδράσουμε. Σας ευχαριστούμε και για το σχέδιο έκθεσης που μόλις λάβαμε. Ίσως προσέξατε πως ε, στην ετήσια έκθεση αναφέρουμε λεπτομερώς το τι συνέβη με την κάθε αναφορά. Στην τελευταία έκθεση για το 2013, στην σελίδα 14 αναφέραμε διάφορα πράγματα που ήταν αντικείμενο αναφορών. και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Πράγματι υπάρχουν τομείς όπου από το μεγάλο αριθμό αναφορών φαίνεται πως ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Λαμβάνουμε πάρα πολλές αναφορές και καταγγελίες από πολίτες όσον αφορά την δικαιοσύνη τώρα. Ένα μικρό σχόλιο για το σχέδιο έκθεσής σας αναφέρεται συγκεκριμένα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ναι βεβαίως κοιτάμε το κεκτημένο και υπό αυτό το πρίσμα εξετάζουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε πως η Κομισιόν ω θεματοφύλακα των συνθήκων πρέπει να εξετάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και το κατά πόσον αυτό μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο και αν μεταφέρει και, και θεμελιώδη δικαιώματα, εξετάζουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Καλωσορίζουμε βεβαίω τον αριθμό των οδηγιών. Τα δεν ξέρω αν αξίζουν και συγχαρητήρια. Όσον αφορά τα νούμερα, μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες διορθώσεις. Κοιτάξτε, το εξή συμβαίνει. Το 2013 ανοίξαμε 761 νέες υποθέσεις, ε, διαδικασίες επί παραβάση. Αλλά οι περισσότερες από αυτές ε, έκλεισαν πριν ε, λάβουμε την απόφαση του δικαστηρίου, γιατί συμμορφώθηκαν τα κράτη-μέλη. Και αν συμφωνείτε θα θέλαμε να διορθωθεί αυτό στην έκθεσή σας. Εκτιμούμε επίσης ε, το ότι επενείται το EU Pilot, το EU Pilot το οποίο από το 2008 έχει γίνει πλέον ένα αποτελεσματικό εργαλείο για έναν σωστό διάλογο με τα κράτη-μέλη πριν να ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση και είμαστε γύρω στο 80% όσον αφορά το ποσοστό επίλυσης. Ποικίλει αυτό αυτό κράτος μέλος, ε, τα αναφέρει η έκθεση τι γίνεται σε κάθε κράτος. Τέλος, η συνεργασία με τα κράτη-μέλη ε, αναφέρθηκε είναι κάτι το κρίσιμο γιατί αυτά εφαρμόζουν δεν εφαρμόζει ούτε η Κομισιόν ούτε η Επιτροπή σας και βεβαίω εκφράζουμε κάποιες αμφιβολίες για το εάν ε, είναι διατεθειμένα τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι τέτοιο και βεβαίως Υπάρχουν και διαδικασίε επί παραβάση και αν δεν συμμορφωθούν τα κράτη-πέλη υπάρχει και το δικαστήριο. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας γιατί εσείς δεν έχετε αυτά τα μέσα. Αλλά βεβαίω είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε συζήτηση για το πώς μπορούμε ως Κομισιόν να σας βοηθήσουμε να λάβετε τις πληροφορίες που θέλετε. Τώρα, ως προς αυτό δεν μπορώ να σας δώσω κάποια συμβουλή, αλλά θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και τέλος. Όσον αφορά τη δική μας επαφή μαζί σας, θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Πρέπει να είναι σαφές το εξής. Όταν κοιτάμε μονομενες περιπτώσεις, βεβαίως, ε, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς διαφάνειας. Αλλά προσπαθούμε ναι, στο πλαίσιο αυτό να δώσουμε στο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Εάν μας πείτε ακριβώς τι θέλετε, ευχαρίστως ε, και εμείς να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Τελευταίο που αναφέρεται στην έκθεσή σας πολύ σημαντικό για εμάς είναι τα λεγόμενα εφαρμοστικά σχέδια. Αυτά τα οποία συντάσσουμε δηλαδή για να μην έχουμε προβλήματα αργότερα στην διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής λειτουργεί το σύστημα, αλλά εξαρτάται βεβαίω από το κατά πόσο το υιοθετούν τα κράτη-μέλη. Άμα δεν το υιοθετούν, εμεί μπορούμε να γράφουμε ό,τι θέλουμε, αλλά εάν δεν το δέχονται, τα κράτη-μέλη ε, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά όπως ξέρουμε λειτουργεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πίτερ. Μια ερώτηση έχω. Τα προβλήματα εμείς δεν τα έχουμε με την Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι εδώ. Ε, και όταν ε, τη θέμε, της μιλάμε. Το πρόβλημα είναι με τα κράτη-μέλη. Γιατί ε, περνάει τόσο καιρό μέχρι να λάβουμε μια απάντηση ή να λάβετε εσεί μια απάντηση από τα κράτη-μέλη. Τι, υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, γιατί βεβαίως χρειαζόμαστε και τα... Χρειάζεται και συμμετοχή των κρατών μελών, έτσι. Εμείς απευθυνόμαστε σε εσά και εσείς στα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι παρατραβάει η υπόθεση. Έκτος αν κάνω λάθος είναι σωστή η εντύπωση που έχω. Κύριε Ριβάση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο όσον αφορά την παρέμβαση των κρατών μελών. Αλλά αφού μιλάμε για στοιχεία αριθμητικά, θα ήθελα να ξέρω σε σχέση με τον αριθμό, με τον αριθμό των αναφορών ε, επί πόσων έχει επιληφθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δίνεται στοιχεία. Θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το ποσοστό των υποθέσεων των οποίων έχει επιληφθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη, θα ήταν σημαντικό και εμείς να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία δεν παρέχουν ε, την αναγκαία προσέγγιση. Κατά την εμπειρία μας αναφερθήκατε στην Ισπανία, έτσι. Ποια ήταν η άλλη? Ιταλία. Ιταλία. Αυτό συμπίπτει. Να πω, ε, δεν έκανα καμία ανάλυση, αλλά νομίζω ήταν Ιταλία, Ισπανία και Τσεχία που δεν συνεργάζονται ιδιαίτερα, τέλος πάντων που καθυστερούν. δεν είναι δεν έχω στατιστικά στοιχεία, απλά παρατηρούμε πως υπάρχουν διαφορές. Το ερώτημά μου είναι, έχετε κάποια συμφωνία κυρίων ή κυριών για να μπορούμε, ξέρω εγώ και εμείς να απευθυνθούμε στους πρέσβεις και να πούμε ε, περιμένουμε εδώ πέρα στην Επιτροπή Αναφορών ε, Έχουμε, τώρα ας πούμε βάλαμε δύο αναφορές ε, για το Μάιο γιατί δεν είχαμε απάντηση από τα κράτη-μέλη. Έτσι. Δεν είναι σωστό και για τους αναφέροντες. Ε, και είναι και ήδη αρκετά παλιές οι αναφορές. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις σχέσεις μας με τα κράτη-μέλη, Έχουμε συμφωνίες κυρίων με τα κράτη-μέλη όσον αφορά το θέμα αυτό. Πρέπει να απαντούν εντός 70 ημερών, 10 εβδομάδες με άλλα λόγια. Όσον αφορά τα τυπικά και τις επίσημες διαδικασίες, αναμένουμε από τις χώρες να απαντήσουν εντός διμήνου. Από την επιστολή επί σειρά ετών αυτή είναι η καθεστική προσέγγιση. Αν δεν απαντήσουν εντό της περίοδου, ε, δεν μπορούν να απαντήσουν εντό της περίοδου, ζητούν παράταση. Και σε κάποιε περιπτώσεις δίνουμε παράταση ενός μηνός ή δύο μηνών. Δεν μπορεί να είναι περισσότερη παράταση από την αρχική προβλεπόμενη περίοδο. Τώρα ρωτάτε πώς μπορείτε εσείς να επηρεάσετε τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να σας βοηθήσει. Τι κάνουμε. Γίνονται διμερείς συναντήσεις με τα κράτη-μέλη. Με τις χώρες που χρειάζεται κάποια υποστήριξη, κάποια συμβουλές και κάτι παραπάνω. διαβιβάζουμε ένα κατάλληλο μήνυμα στα κάτι μέλη. Η σύμφωνη γνώμη τους δεν είναι κάτι που αφορά εμάς. Πρέπει να σας βοηθήσουμε ίσως για το πώς θα μπορούσατε εσείς να πιέσετε τα κάτι μέλη. Δεν ξέρω αν θα έχει τέτοια εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι διαμεσολαβητής. Έχουμε πολλά καθήκοντα, αλλά δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αυτό. Στοιχεία explain to you that we had... Να σας εξηγήσω. 2013. 761 διαδικασίες κατά παράδοση ξεκίνησαν κατά των 100 μελών και 731 ποιο είναι το ποσοστό περίπου 90% έκλεισαν οι διαδικασίες πριν βγει απόφαση του δικαστηρίου. Αυτά είναι τα γενικά στοιχεία για το 2013. Για τις αναφορές ομολογώ ότι δεν διαθέτουμε τα στοιχεία, τα έχουμε εδώ. Αλλά πιστεύω ότι αφορά τις καταγγελίες εν γέννη και δεν υπάρχει πραγματική διαφορά μεταξύ καταγγελιών που περνούν από την Επιτροπή Αναφορών και εκείνων που υποβάλλονται απευθεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα αναμένω ότι το ποσοστό επιλύσεως των προβλημάτων είναι περίπου 10% και παραμένει το ίδιο. Το 10% είναι υποθέσεις εκείνες όπου τελικά καταλήξαμε στη δικαστική απόφαση. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης την εξέλιξη. Δεν είμαστε μόνο θεματοφύλακα τη συνθήκη σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είμαστε και εκτελεστέ των δικαστικών αποφάσεων. Αυτό πιο σοβαρό. Και μπορούμε να επιβάλλουμε και οικονομικέ κυρώσει όταν διώκονται κάτι μελη για μη εκτέλεση αποφάσεων δικαστικών. Ελπίζω όλα αυτά να σας διαφωτίζουν. Πολύ καλά. Ορίστε. Αυτό σημαίνει ότι 761 αναφορές, οι 731 μπόρεσαν να διεκπεριωθούν, άρα μένουν 30 αναφορές που οδηγούνται τελικά σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό, αυτό σημαίνει αυτό που είπατε. Εστέ πιο σαφής. Μιλάμε για 10%. Ποιο είναι το στοιχείο. Θα προσπαθήσω γαλλιστή. Είχαμε 760 761 διαδικασίες κατά των κρατών μελών, κατά των 28 κρατών μελών. Άρα, στείλαμε επιστολή, επιστολές προειδοποίησης, αιτιολογημένες επιστολές και προσεφήγαμε και στο δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, σε κάποιες, κάποιες υποθέσεις επελήφθησαν διότι δέχτηκαν τα κρατημένα κάνουν αυτό που έπρεπε. Αποτέλεσμα. 31 θαρώ, 31, 32 υποθέσεις αποφάσισε το δικαστήριο. 10% δηλαδή από όλε τις υποθέσεις που ξεκινήσαμε διαδικασίες παράβασης κατά αυτόν το δικαστήριο αποφάσισε και μετά εκτελέστηκε απόφαση του δικαστηρίου από τα κράτη-μέλη με, καμιά φορά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι παρακολουθεί αυτή η περιπτώση πολύ προσεκτικά τις αποφάσεις και πώς εκτελούνται οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να σας απάντησα. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέχρι 30 Μαρτίου υποβολή τροπολογιών, ψηφοφορία στην Επιτροπή Αναφορών προβλέπεται για 5 Μαΐου και στην στις 6 μέχρι 9 Ιουλίου του 2015. Ε, πάμε στους αναφέροντες, στο σημείο 8, πάμε στην αναφορά 1932 Πολ Λάγκεν όσον αφορά τις ε, νοσοκομιακές δαπάνες ε, και πώς καλύπτονται αυτές σε περίπτωση μεταφοράς, μετάβασης άλλο κράτος μέλος ακύρωση ασφαλιστηρίου συμβολίου υγεία για κάλυψη νοσοκομιακών δαπανών σε περίπτωση μετακόμιση άλλο μέρα. Ε, η Ελεονόρα θέλει κάτι να πει. Συγγνώμη, ήθελα να παρέμβω όχι από αυτού, αλλά από του προηγουμένου τη Προέδρου για την ανακοίνωση τη Ακροάσεω για την αναφορά για το Vivisection. Λοιπόν, σαν μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ζητήσαμε μέσω του συντονιστούς να συμμετάσχει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά το θέμα αυτό για να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, το vivisection, γιατί θα πρέπει να έχουμε και τη ε, συμμετοχή της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται μόνο για την ευημερία των ζώων σαν θέμα, αλλά και για την υγεία. Άρα είναι σημαντικό ε, για τους ευρωπαϊκούς πολίτες. Ήθελα να ζητήσω από εσά αν μάθατε αν θα συμμετάσχει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό. Hm? Λοιπόν, καλώς. Ε, θα συμμετάσχει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα κάνουμε τα δέοντα. Πάμε λοιπόν σε αυτή την αναφορά του κυρίου Πολ Μάγκεν, που είναι στο σημείο 8 της μέσης διάταξης. Οι αναφέροντες απουσιάζουν. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Λούκα Πορτέλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατανοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προβλήματα των αναφερόντων, του αναφέροντος. Λάβαμε καταγγελίες από πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως για παρόμοιο θέμα και αξιολογούμε κατά πόσο και πώς και πότε μπορούμε να βελτιώσουμε ε, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με το θέμα. Το θέμα είναι ότι η νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ενώσεω βασίζεται επί δύο αρχών. Την αρχή της τοποθεσίας των ασφαλιστικών κινδύνων και τη ελευθερία της συνάψεω συμβάσεων. Η πρώτη αρχή, η αρχή του τόπου ε, του ασφαλιστικού κινδύνου, τι σημαίνει. Ότι ένας καταναλωτής μπορεί να ασφαλιστεί από ασφαλιστική εταιρεία η οποία έχει αδειοδοτηθεί στο κράτος μέλος της χώρας που κατοικεί ή από ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα κατοικία του από το εξωτερικό σύμφωνα τη ελευθερία των συνθήκων. Η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν υποχρεώνει τι ασφαλιστικέ εταιρείε να είναι ενεργέ σε όλα τα κράτη-μέλη. Η δεύτερη αρχή είναι η αρχή τη ελευθερία τη σύμβαση, τη σύναψη σύμβαση. Σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείε και οι καταναλωτές μπορούν να συμφωνήσουν και να συνάψουν διάφορες ασφαλίσεις υπό διάφορους όρους και το γραφικό πεδίο κάλυψης και μπορεί να αποφασίσουν να αποκλείσουν τα παρεχόμενα ωφέλη από την ασφαλιστική εταιρεία που θα παρέχονται σε άλλο κάτω μέλος. Τώρα, όπως είπα, αξιολογούμε ενδεχόμενες βελτιώσεις. Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα. Το παράδειγμα τις οδηγίες για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων που καλύπτει τις, ασφα... τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις τρίτων μερών ευθυνών. Η οδηγία βασίζεται επί, της... επί του ενίου ασφαλίστρου και της ειδικής αρχής. Άρα ο οδηγός ασφαλίζεται από την ασφαλιστική του εταιρεία και όποτε προξενεί σε άλλο κάτω μέρο το εξωτερικό ατύχημα, εγγυάται η ασφάλισή του ότι θα παρέχονται ωφέλη στο άλλο κράτος μέλος. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να βρούμε παρόμοιες ή ανάλογες λύσεις στον τομέα σε άλλες ασφαλιστικές, ε, σε ασφαλιστικούς τομείς όπως είναι η ιατρική ασφάλιση που αναφέρει και ο αναφέρον. Αυτά και ευχαριστώ. Στους άλλους από τους συντονιστές ε, ήθελε το λόγο πείτε. Ja, jetzt, ähm, <clears throat> die Frage geht jetzt fast an meine Kollegen im Ausschuss, weil äh, Κοιτάξτε. Λάβαμε μία ενδιαφέρουσα απάντηση της Κομισιόν. Παραπονείται κάποιος εδώ πέρα για την ασφάλιση και βεβαίως εδώ πέρα κινδυνεύει στην ασφάλιση υγείας η εσωτερική αγορά. γιατί βρίσκεται εδώ πέρα ένας άνθρωπος από ένα κράτος μέλος και ανακαλύπτει ότι δεν είναι πλέον εγγυημένη η κάλυψή του και απειλείται με τεράστια επιπρόσθετα ασφάλιστρα. Η Κομισιόν λέει πως είναι πρόβλημα. Έχουμε το παράδειγμα των αυτοκινήτων, όπου η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει αυτομάτως πανευρωπαϊκά. Οπότε εδώ πέρα τι γίνεται ε, αφενός λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί η κατάσταση είναι αυτή που είναι, αλλά η Κομισιόν λέει πως πρέπει να γίνει κάτι. Ε, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Και το ερώτημα λοιπόν είναι τι κάνουμε τώρα. Το κλείνουμε, συμπεριλαμβάνουμε και την ε, αρμόδια επιτροπή. Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τι να πω. Alguna intervención más? Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Ωραία. Ε, λοιπόν, υπάρχει μια πρόταση του Πίτερ, αλλά φαίνεται πως και η Κομισιόν λέει πως αξιολογεί την εφαρμογή της ε, οδηγίας. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση λοιπόν όσο περιμένουμε την αξιολόγηση της Κομισιόν να το αφήσουμε ανοιχτό το θέμα. Γιατί περιμένουμε κάποια συμπεράσματα από την Κομισιόν για την εφαρμογή. Συμφωνείτε? Ωραία. Αποφασίστηκε. Λοιπόν, περνάμε στο 9 και 10 να... που ζητήθηκε να πάνε μαζί αυτά. 8-9 αφορά διάφορες αναφορές και αναφέρονται σε 1635 για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και τις σχετικές εισαγωγές τροφίμων. Ένα άλλο, ε, μια άλλη αναφορά είναι η 1960 για την αναστολή διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ για τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. Μετά η ε, 27-21 για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών η 28-59 με 120 υπογραφές σχετικά με την ΤΑΦΤΑ και άλλες 26 αναφορές και βεβαίως ε, έχουμε και την γνωμοδότηση μετά για τις διαπραγματεύσεις. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα ένας αναφέρον παρόν ο Μπρούνο Κραμ και θα ήθελα να του δώσω τον λόγο και μετά συνεχίζουμε. Έχετε τον λόγο. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, όταν κατέθεσα την αναφορά μου το 2013, η συμφωνία αυτή δεν ήταν πάρα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Χωρίς την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών τα τελευταία χρόνια, το ίδιο θα συνέβαινε και σήμερα. Η συμφωνία αυτή έγινε όπως και στο παρελθόν χωρίς συμμετοχή του κοινού. Οι επιθυμίες των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων ήταν σημαντικότερες. Όμως πλέον χάρη στο ίντερνετ έχει αυξηθεί πάρα πολύ η απέτηση των πολιτών για συμμετοχή και έτσι νομίζω συγκινήθηκαν οι Βρυξέλλες και το Κοινοβούλιο. Και στις δύο του Ατλαντικού ζητάνε οι πολίτες συμμετοχή και διαφάνεια όταν μικρές ελίτ αποφασίζουν το μέλλον τους. Η ανάγκη αυτή των ανθρώπων και στις δύο όχθες του Ατλαντικού ε, πέφτει σε ένα παγκόσμιο κενό γιατί οι πολίτες μέχρι στιγμής δεν είχαν καθόλου επιρροή στους κανόνες του παιχνιδιού. Ο καπιταλισμός μπορεί μέχρι στιγμής να κατάφερε να ξεπεράσει τις ρυθμίσεις του ε, και σε παγκόσμιο επίπεδο ισχύει από ό,τι βλέπουμε το δίκαιο του ισχυρότερου. Εάν το διεθνές δίκαιο είναι πάνω από το εθνικό όπως στην TTIP τότε ζητάνε οι πολίτες το αυτονόητο δικαίωμα στην συναπόφαση και όμως πολύ περισσότερο από αυτό ζητάμε διαφάνεια έχουμε το ανθρώπινο δικαίωμα να δούμε τα διαπραγματευτικά έγγραφα όταν παρεμβαίνουν τόσο πολύ στην δημοκρατία όσο η TTIP. Δεν ξέρουμε πλέον οι πολίτες τόσο πολλά όσο ξέρουν οι λομπίστες και οι βουλευτές μας. Η TTIP συμπεριλαμβάνει προστασία των καταναλωτών, τρόφιμα, συντάξεις, νερό, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, όλους τους τομείς της ζωής και το ερώτημα είναι εάν θα ρυθμιστούν όλα αυτά προς όφελος των μεγάλων εταιριών χωρίς να έχουν λόγο οι άνθρωποι, αυτοί, οι της Ευρώπης και του κόσμου. Από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά η ευθύνη και η διοίκηση φεύγει από τα δημοκρατικά κοινοβούλια και πηγαίνει στις εταιρείες. Θα μπορούσαμε να έχουμε Επίσης, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μια λεγόμενη ζωντανή συμφωνία, η οποία δηλαδή θα αναθεωρείται συνεχώς και κατά της οποίας δεν θα μπορεί να προσφύγει κανείς. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εάν θα έχουν οι εταιρείε περισσότερα δικαιώματα από τις δημοκρατίες για να εκβιάζουν σε αδιαφανή διαιτητικά δικαστήρια. Θα πρέπει λοιπόν Επιτέλους να σταματήσουμε τις εταιρείε. Δεν είναι δυνατόν τα παγκόσμια προβλήματα να λύνονται χωρίς συμμετοχή των ανθρώπων που ζουν στον κόσμο αυτόν. Το θέμα είναι εάν θα συνεχίσουμε με την προστασία των ε, δικαιωμάτων αυτών του εμπορίου να καταστρέφουμε τις φτωχότερε χώρες και το εάν Θέλουμε έτσι με αυτό τον ε, τρόπο να πουλάσουμε ακόμα και την ιδιωτική σφαίρα του πολίτη. Ο πολίτης της δημοκρατίας μας πρέπει επιγόντως να αποκτήσει το δικαίωμα να μάθει τα πάντα. Και δεν θέλουμε μόνο διαφάνεια, θέλουμε και συναπόφαση. Γιατί η συμφωνία αυτή αφορά το μέλλον των δημοκρατιών μας. Η έλλειψη διαφάνειας είναι αυτό το οποίο συνδέει όλη αυτή την υπόθεση. Είναι ένα σύμπτωμα της, ενός μοιραίου λάθους το οποίο θα συνεχιστεί με τα διαιτητικά δικαστήρια. Εμείς πιστεύουμε στη δημοκρατία, πιστεύουμε στην ποικιλομορφία της Ευρώπης. Ελπίζουμε λοιπόν οι βουλευτές να μην υπογράψουν μια συμφωνία την οποία δεν γνωρίζουν εις βάθος και δεν συναποφασίζουν ενώστε την φωνή σας μαζί μου. Δεν είναι δυνατόν να λέτε μόνο ναι ή όχι. Δεν είναι δυνατόν να σας αρκεί αυτό ως ε, δημοκράτες. Δεν είναι διαφάνεια αυτό το πράγμα. Πείτε όχι στην TTIP και είπε ναι στην διαφάνεια, τη συμμετοχή και την δημοκρατία για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός μικροφώνου Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε τον κύριο Κράμε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω διότι ε, μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε στη σημερινή συνεδρίαση και να διαλευκάνουμε ε, κάποια στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Κράμ στην αναφορά του. Τα δύο βασικά που θίγει ο κύριος Κράμ είναι η διαφάνεια ή κάτι που αντιλαμβάνεται εκείνος ως έλλειψη διαφάνειας και δεύτερον ότι θα υποβαθμιστούν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω της TTIP. Εγώ προσωπικά είμαι αρμόδιος για τη διαπραγμάτευση των, ε, της υγειονομικής και φυτογειονομικής στοιχής ε, της TTIP. Ασχολούμαστε λοιπόν με τα πρότυπα και τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υπερασπιστούμε και στις διαπραγματεύσεις για την TTIP. Θα ήθελα αρχικά να επαναλάβω αυτά που συμπεριλάβαμε στην απάντηση που στείλαμε για την αναφορά ότι δεν ε, εγκυμονεί η διαπραγμάτευση κανένα κίνδυνο υποβάθμιση των υψηλών προτύπων ασφαλείας για την ασφάλεια των τροφίμων. Θέλω όμως να στοιχειοθετήσω αυτή την ε, απάντηση. Από το σχέδιο απάντησης έχουν συμβεί πολλά πράγματα, έχουν συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια προηγουμένου άσκηση ε, διαφάνειας ε, για το κείμενο των διαπραγματεύσεων, για αυτό το κεφάλαιο και για άλλα και έκτοτε έχουν δημοσιευθεί μετά από πρωτοβουλία της Επιτρόπου Μάλμστρομ αυτά τα σχέδια στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο κοινό. Ο Σκράμ, οποιοδήποτε στον κόσμο μπορεί να δει το ε, κείμενο που διαπραγματευόμαστε για το κεφάλαιο για τα φυτογενομικά και γενομικά μέτρα αλλά και για όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια. Οι συνάδελφοι θα συζητήσουν θα σας παρουσιάσω το ζήτημα της διαφάνειας με περισσότερες λεπτομέρειες, όμως ήθελα να ξέρω, να γνωρίζετε μάλλον ότι υπάρχει η διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαπραγματευτική θέση ε, των Αμερικανικών αρχών σε ειδική αίθουσα ανάγνωσης. Βλέπετε λοιπόν πως η προσέγγιση που υιοθετούμε σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των προτύπων. Το αντίθετο είναι ευκαιρία για τον αγροδιατροφικό τομέα. Σε όλα τα επίπεδα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συναρμόδιοι επίτροποι ακολουθούν αυτή την αρχή ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμα τα πρότυπα ασφαλείας των τροφίμων. η μη χρήση των ορμονών για την ε, ε παραγωγή, η χρήση αντιβιωτικών για τα ε, ε, προϊόντα ζώων και οι κανόνες για τη βιοτεχνολογία θα διαφυλαχθούν. Αυτή την αρχή την προσυπογράφουν και οι Αμερικανικές αρχές. Βάσει των υποχρεώσεων που έχουν και δύο πλευρές στα πλαίσια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου επιφυλάσσεται το δικαίωμα να εξασφαλίσουν ε, την κατοχήρωση των προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων και οι δύο πλευρές. Ε, χαιρόμαστε που είχαμε όμως αυτή την ε, ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με την Κοινωνία των Πολιτών και την ε, Επιτροπή Αναφορών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπαθούμε έτσι να διασκεδάσουμε οποιασδήποτε ανησυχίες υπάρχουν για την υποβάθμιση των υψηλών προτύπων ασφάλειας των τροφίμων. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Ο κύριο Λούτσε Λίνκερ θέλει να παρέμβει από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα προσθέσω κι εγώ κάποιε παρατηρήσεις. Αυτές οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε μια διαπραγματευτική εντολή που έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη. Ε, έχει δημοσιευθεί στο μεταξύ διαπραγματευτική εντολή και αυτό ε, η ρίστον παρόδο ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι δημόσια η διαπραγματευτική εντολή. Όποιος πολίτης το επιθυμεί μπορεί να δει μέσα στην εντολή ποιες είναι οι κατευθυντήρες γραμμές για τις διαπραγματεύσεις. Ε, για να ε, γίνει κατανοητό τι πρέπει και τι δεν πρέπει να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποβάθμιση των προτύπων δεν εντάσσεται στη διαπραγματευτική εντολή και είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμες οι αρχές, ούτως ή άλλως δεν είναι να το κάνουμε. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Κάμ και συμφωνώ γιατί γνωριζόμαστε και καλά με τον κ. Κάμ, Ε, αναφέρει, ε, ε, αυτά που αναφέρει λοιπόν δεν στοιχειοθετούν βάσει διαπραγματευτική διαπραγματευτικής Ε, σε σχέση τώρα με προηγούμενε εμπορικέ διαπραγματεύσεις θα έλεγα ότι είναι η βάση στην οποία ε, δράζονται οι πραγματεύσεις για το TTIP. Δηλαδή 50 χρόνια διμερών συμφωνιών ε, ελευθέρου εμπορίου με την Κορέα παραδείγματο χάρη διαπραγματεύσεις μόλις ολοκληρώσαμε με τον Καναδά. Ε, το κείμενο υπάρχει στο διαδίκτυο, όλοι μπορούν να το συμβουλευτούν και να δουν το περιεχόμενό του. 50 χρόνια εμπειρίας λοιπόν και επίσης συνεχίζεται διαπραγματεύση Δεν έχουν ολοκληρωθεί και για τη διαφάνεια, όπως είπε και ο κύριος Ένση, είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ το θέμα της διαφάνειας και για τη, ειδικότερα για την Επίτροπο Αρμόδια για το Διεθνές Εμπόριο, την κυρία Μάλμστρομ. Ε, στη πλήθεια της ΤΤΙΠ εκδόθηκε και ανακοίνωση σχετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια σειρά από βήματα που έχει ήδη αναλάβει και θα ε, αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλιστεί ε, ακόμη ευρύτερη διαφάνεια Στι 7 Ιανουαρίου, μετά από εφαρμογή αυτή τη ανακοίνωση, άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύει όλα τα διαπραγματευτικά έγγραφα, όπω είπε και ο συνάδελφο μόλι τώρα, στο διαδίκτυο είναι ανευπροηγουμένο αυτό το βήμα στα, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλες παρελθούσες διαπραγματεύσεις ε, με οποιοδήποτε εταίρο. Εξηγούμε με σαφήνεια το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, το στόχο που επιδιώκουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις και όπως είπε ο συνάδελφος, είναι ξεκάθαρα πλέον τα τεκμήρια. Επίσης δημοσιεύουμε τα έγγραφα που ε, αποστέλουμε στο Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη, ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους τους πολίτες, να ξέρουν ακριβώς τι στέλνουμε στους προσώπους τους. Ε, είναι ε, η ιστοσελίδα μας επίσης ε, λεπτομερέστατη με πληροφορίες επεξηγηματικές πέραν από τα διαπραγματευτικά έγγραφα για τους μη ειδικού και επίσης εκατοντάδες πολίτες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή ως ενημερωτικές συσκέψεις πριν και μετά τις διαπραγματεύσεις υπάρχουν συσκέψεις, υπάρχει και μια διαπραγματευτική Ομάδα που λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2013 που μετέχουν εκπροσώποι της κοινωνίας των πολιτών και ε, συζητούνται ζητήματα ε, που ενδιαφέρουν την κοινωνία των πολιτών. και πιο σημαντικό είναι ε, ότι ακολουθούμε την πολιτική της ανοιχτής πόρτα. Δεν υπάρχει προτιμησιακή πρόσβαση σε οποιαδήποτε ομάδα επιχειρηματική ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανθρώπων. Όλοι έχουν ισότιμη πρόσβαση τα έγγραφα και τι πληροφορίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να και κάποια άλλα ζητήματα που ανέφερε ο κ. Σκράμι, η νομοθετική συνεργασία με το Συμβούλιο, στην οποία αναφέρθηκε, είναι μέρο τη πρότασή μα για την ε, ε, κανονιστική συνεργασία στα πλαίσια τη TTIP. Υπάρχει ε, το διαπραγματευτικό κείμενο που δημοσιεύσαμε, μπορείτε να το συμβουλευτείτε για να δείτε ότι προτείνουμε ένα φόρουμ συνεργασίας, ε, κανονιστική συνεργασίας ε, με τις ΙΠΑ, που ξεκάθαρα δεν έχει καμία αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για φόρουμ βήμα συνεργασίας. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, για το ζήτημα της ε, προστασίας των επενδυτών και του μηχανισμού ρύθμισης διαφορών κράτους επενδυτή. Δεν θα πω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά παραπέμπω στη σύσκεψη των συναδέλφων σας από την Επιτροπή Ήτρια που θα λάβει χώρα αύριο και αυτό είναι ένα από τα σημεία της της διάταξης, συζήτηση μετά από έτοιμα της κυρίας Μάνστρομ όπου βλέπουμε ε, ότι στο κεφάλαιο της προστασίας των επενδυτών θα αναδειχθεί σε μία από τις βασικότερες προτεραιότητες στο θέμα δηλαδή της διεύθυνσης των διαφορών κράτους επενδυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές. Θα ξεκινήσω τον κύριο Βαλέσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Ευχαριστώ κύριε Κάμπ που είστε εδώ παρόν. Προσωπικά ήλπιζα ότι θα έχουμε πολλούς περισσότερους αναφέροντες παρόντες διότι λάβαμε περίπου 30 αναφορές όσον αφορά διαφορετικά θέματα, αλλά χαίρομαι που είστε εδώ μαζί μας, διότι προφανώς θίγεται ένα σημαντικότατο σημείο. Τις τελευταίες εβδομάδες συμμετείχα σε διάφορες συναντήσεις επί του θέματος με διάφορους συντάκτες σε όλες τις γνωμοδοτικές επιτροπές διότι φαίνεται σχεδόν ότι κάθε επιτροπή του Κοινοβουλίου θα γνωμοδοτήσει επί του TTIP. Εστέ βέβαιος λοιπόν ότι εργαζόμαστε σκληρά για να καλύψουμε όλες αυτές τις καταγγελίες και ανησυχίες, διότι προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε παρούσες όλες τις πληροφορίες, ούτως ώστε να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση κι εσείς. Το θέμα σας δεν είναι το μόνο που πρέπει να εξετάσουμε οι αναφορές που λαμβάνουμε, που λάβαμε μάλλον, κάλυψαν θέματα που αφορούσαν την ποιότητα των τροφίμων, ε, την ψηφιακή αυτοδιάθεση, τη διαφάνεια, ε, οικονομικό αντίκτυπο, το ISTS, ε, Άρα υπάρχουν πολλά θέματα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε δύο ζωτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιγράφονται στις διαπραγματεύσεις TTIP. Πρώτα απ' όλα Θέλουμε να πετύχουμε μια εμπορική συμφωνία ισορροπημένη και λογική μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ, να εξαλείψουμε μετά του θελωνιακού δασμού και να σημειώσουμε πρόοδο προ αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων για τα προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ. Αυτά υφίστανται σαν στόχοι γενικότερα και σημαντικότερο στην ενακτή διαδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ίδιος, κατέστησε σαφέστατο ότι η Ευρώπη δεν θα θυσιάσει την ασφάλεια, την υγεία, την προστασία την κοινωνική και την προστασία των δεδομένων, τις σχετικές προδιαγραφές και την πολιτισμική μας ποικιλομορφία στις διαπραγματεύσεις. Για εκείνον η ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία των προσωπικών στοιχείων των Ευρωπαίων θα είναι μη διαπραγματεύσιμα. Υπάρχει αυτό και το έχουμε μπροστά μας, το έχω. Παρατηρήσαμε τις τελευταίους μήνες όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα στα πλαίσια πνεύματος διαφάνειας και αμοιβές εμπιστοσύνης υπό το φως της παρούσης συζητήσεως βλέπουμε ότι ισχύει και αυτό και εδώ και βλέπουμε ότι τα σημαντικότερα θέματα όπως οι ορμόνες, το ο κρέας και η νομοθεσία για τους γενετικά τοποποιημένους οργανισμούς είναι θέματα που συζητούνται και θα πολεμήσουμε ούτω ώστε να παράσχουμε τη σωστή ασφάλεια και τα σωστά, σωστές προδιαγραφές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμιά φορά απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, μας ενημερώνει και θεωρώ ότι είναι οι διαφανέστερες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Προφανώς θα προσέξουμε και το υπόλοιπο των διαπραγματεύσεων, αλλά τα περισσότερα θέματα ε, με ικανοποίησαν το πώς εκαλύφθησαν. Θα ετοιμάσω ή μάλλον ετοίμασα τη γνωμοδότησή μου και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι θα συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα θέματα και θα ήθελα να ζητήσω τις άλλες πολιτικές ομάδες, τους άλλους συντονιστές να μου στείλουν τα ονόματα των σκιωδών εισηγητών, ούτως ώστε να μπορέσω να προγραμματίσω συνάντηση, ελπίζω πριν από τις πασχαλινές διακοπές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε εκτενώς την γνωμοδότηση και να μπορέσουμε όλοι να ικανοποιηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που είστε παρόν, κύριε Κάμ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Βαλέσα. Ο κύριος Ρέντα, η κυρία Ρέντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ε, παρουσίαση αυτή της αναφοράς για το θέμα της TTIP. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα ανοιχτά με την Κομισιόν. Πρέπει να πω πως κάποιες από τις παρατηρήσεις της ε, Κομισιόν ε, μπαίνουν στην ουσία, αλλά κάποιες ε, την προσπερνούν. Το θέμα εδώ πέρα δεν είναι το ότι υπάρχει ανησυχία ότι υπάρχουν υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κινδυνεύει η εμπορική συμφωνία, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες ανησυχίες για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον να ε, μπορεί να εγκρίνει από μόνη της ε, κανονισμούς. Ε, έχουμε ακρόαση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ακριβώς για το θέμα αυτό και το ISTS όπου υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές αμφιβολίες για το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. για τα νέα προβλήματα και παιδεία πολιτικής που ζητάνε ρύθμιση και να δούμε το τι θα γίνει αν θα διατηρηθούν όλα αυτά εάν εγκριθεί η, η δημοσιοποίηση της διαπραγματευτικής εντολής είναι οπωσδήποτε ένα σωστό βήμα ε, και οπωσδήποτε χαιρέτησε η ομάδα μου τώρα εάν εντωμεταξύ υπάρχουν και άλλα διαπραγματευτικά κείμενα τα οποία δημοσιεύτηκαν είναι οπωσδήποτε κάτι το σημαντικό και διατηρείται έτσι η πίεση στους Αμερικανούς να δημοσιοποιηθεί όλη η διαπραγματευτική διαδικασία. Γιατί πράγματι ο κόσμος είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος. τώρα ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι αδιαφανείς δεν ξέρω αν ισχύει ως δικαιολογία. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο οπωσδήποτε και η Κομισιόν να λάβουν υπόψη το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς κόσμου. Ευχαριστώ. Η κυρία Ριβάζη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσαμε καταρχάς για διαφάνεια. Μιλάτε για τι πράγματα, ναι. τι εννοείτε. Λέτε ότι οι συντονιστέ μπορούν να έχουν πρόσβαση στι διαπραγματεύσει και στα ενοποιημένα κείμενα. Δεν μπορούν να κάνουν όμω φωταντίγραφα, δεν μπορούν να πάρουν φωτογραφίε, δεν μπορούν να κρατήσουν σημειώσει. Το αποκαλείτε αυτό διαφάνεια. Ε, έχετε μια μικρή. Ε, να ρίξω μια ματιά, αλλά δεν επιτρέπονται φωτοαντίγραφα. Αυτή είναι η διαφάνεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις ενώσεις, τα συνδικάτα δεν μπορούν να έρθουν Και όλοι οι βουλευτές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση. Εγώ που ενδιαφέρομαι για την υγεία δεν μπορώ να έχω πρόσβαση. Θα πρέπει να περάσω μέσω συντονιστού και ο συντονιστής δεν ξέρει τι είναι ενδιαφέρον και δεν μπορεί σε αυτά που τον ενδιαφέρουν να πάρει φωτοτυπίες. Αυτή είναι η διαφάνειά σας. Να σας πω αυτή τη στιγμή εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζετε κατά της Ευρώπης. Διότι εμεί όταν είμαστε επιτόπου πρέπει να εξηγήσουμε μετά στου πολίτε μα και να πούμε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι ακόμα και οι ενώσει δεν μπορούν να γνωρίζουν ακριβώ τι γίνεται με τι διαπραγματεύσει, πώ μπορούμε να υπερασπιστούμε την Ευρώπη. Μετά λέτε θα εναρμονίσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τίθεται θέμα να αμφισβητηθεί η νομοθεσία ρίτς, τι κάνουμε του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού, η τικηταθεσία κλπ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν, είμαστε, δεν κινούμαστε από των ιδίων αρχών. Στην Ευρώπη ασχολούμαστε στην αρχή της πρόληψης, κινούμαστε βάση αυτή. Κάθε μόριο που εξέρχεται γίνεται υγειονομική περιβαλλοντική μελέτη. Αλλά είπα δεν κάνουν τίποτα από αυτού. Όλα τα μόρια ε, βγαίνουν στο περιβάλλον και χρειάζεται ε, κίνδυνος για να εξαλειφθούν. Έχουμε εντελώ διαφορετικό τρόπο να κινούμεθα. Κάντε να δεχτούν οι Αμερικανοί την αρχή τη πρόληψη και την αυτή περιπτώση μπορούμε να συζητήσουμε. Γιατί και τα θεσία όσον αφορά του γενετικά τροπημένου οργανισμού. Στην Αμερική υπάρχουν παντού οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και μολύνουν τα γειτονικά, τι γειτονικέ εκμεταλλεύσει. Πώ θα επιβάλλουμε στι ΗΠΑ ότι τα τρόφιμα που θα εισάγουμε θα έχουν την ετικετοθεσία όσον αφορά του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Έχουμε εντελώ διαφορετικού τρόπου εργασία και διαβάζω αυτό που λέτε όσον αφορά την διατροφική υγιεινή Στη ΣΥΠΑ, αν ε, έχουν τα χλωριωμένα ε, κοτόπουλα και ακτινοβολούν τα τρόφιμα. Ξέρετε την ακτινοβολία, είδα ένα ρεπορτάζ πρόσφατα. Το βόλιο κρέας, το στέικ, δεν έχουν την πρόληψη όπως στην Ευρώπη στη ΣΥΠΑ. Σαν τελευταία προσβυγή ακτινοβολούν για να εξολοθέψουν τα μικρόβια. Εμείς δεν έχουμε καθόλου αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και λέτε ότι καμία συνθήκη κατά των μικροβίων δεν θα εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν αποδειχτεί επιστημονικά ότι προσφέρει ωφέλη στους καταναλωτές. Ποιος θα το κάνει αυτό, η ΕΦΣΑ. Και ξέρετε ότι τώρα βλέπουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας η ακτινοβολία. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να έχει γίνει από αυτού. Όμως, και διαρωτώ με, σε ποιο κόσμο θα μας βάλετε όσον αφορά την επιστημιστική ασφάλεια, την ασφάλεια των τροφίμων, εγώ όσον αφορά το θέμα, τι να πω, όσον αφορά τα φάρμακα μετά. Εγώ ε, βλέπουμε τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τους ε, Καναδούς. Τι κάνουμε όμως. Ε, τα φαρμακευτικά εργαστήρια επιβάλλουμε να παρατείνουμε τη διάρκεια των, των φαρμάκων διότι δεν είναι γενώσιμα. Εμείς τι κερδίσαμε. Εμείς πολεμάμε να υπάρχουν γενώσιμα. Αλλά τα φαρμακευτικά εργαστήρια θέλουν να παρατείνουν, να καθυστερήσουν διότι δεν έχουν την ίδια νομοθεσία οι Όταν βλέπω αυτά και όταν βλέπω τη συμφωνία σε επίπεδο αλένα, δεν ξέρω τι θα μας δώσει η συμφωνία. Θα ενθαρρύνει το εμπόριο στο επίπεδο των μεγάλων λόμπι και οι ρυθμίσεις και ο τρόπος λειτουργίας των Αμερικανών δεν είναι ο ίδιος όπως ο ευρωπαϊκός. Ε, μετά το STS ε, γίνονται διαβουλεύσεις 150 χιλιάδες απαντήσεις όσον αφορά τη διαβούλευση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γνωρίζει όλα αυτά και λέει υπήρξαν πολλές παρόμοιες απαντήσεις, δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Βλέπετε τι εικόνα στέλνει αυτό, τι δημιουργεί. Μας λέτε ότι οι βουλευτές δεν εξυπηρετούσε τίποτα. Είναι άρνηση της πολιτικής εξουσίας αυτή. Και το ISDS έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Είδαμε ότι τα εργαστήρια είτε της πετρελαϊκής βιομηχανίας ή άλλα εργαστήρια φαρμακοβιομηχανίας επετέθησαν κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων. Διότι έχουμε μια νομοθεσία που επιτρέπει πρόσβαση στις κλινικές δοκιμασίες. Τα, τι έκαναν τα φαρμακευτικά εργαστήρια, επετρεψαν κατά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων ή είπαν ότι είναι μυστικό, επαγγελματικό αυτό κλπ. Αυτό τον κόσμο θέλετε να οικοδομήσουμε μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο και αν είναι για να πάμε αντίθετα, εγώ λέω που είναι στη Γαλλία, ψηφίσαμε ένα νόμο για την απαγόρευση ε, την υδρολογμάτωση. Αλλά μετά έγινε επίθεση κατά της Γαλλίας μια εταιρεία, ε, τις δικαστές θα πούνε ποιε οι αποζημιώσεις πρέπει να πληρώσει η Γαλλία όσον αφορά αυτή την απόφαση. Αλλά είναι άρνηση κάθε πολιτικής ε, δύναμη σε επίπεδο Ένωση και 100 μελών. Τα κράτη-μέλη σα έδωσαν μια εντολή. Πράγματι, αληθεύει αυτό. Και τώρα επιτίθεστε κατά των κρατών μελών, ούτω ώστε ακριβώ να, ε, να αρνηθούν τελικά το TTIP. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα τα κράτη-μέλη και ο πολίτη Ευρωπαίο. Είδατε την άνοδο του Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία που ασχολήθηκε και εκμεταλλεύτηκε το TTIP και είπε δεν θα υπάρξει πλέον προστασία. Δεν μα λέτε αυτό στο κείμενο. Θα λέτε ότι θα υποχρώσετε τι ΗΠΑ να έχουν πιο περιοριστική νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Ρίμπαση. Ελεονόρα, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσία εδώ του αναφέροντος. Εγώ ήθελα να επιθυμίσω ότι αυτές οι πολυάριθμες αναφορές που λάβουμε αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες των πολιτών και ήθελα να ότι υπάρχει έγινε μια απόπειρα μάλλον πρωτοβουλία ε, πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών που απερίφθη όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σημαντικό να το υπενθυμίσουμε, όμως συνεχίζεται ακόμα η εκστρατεία και μαζεύτηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές, άρα το θέμα είναι σημαντικό και πρέπει να εισακουστούν τα αιτήματα που γίνονται από πλευρά πολιτών. Και διότι αυτή η συνθήκη μας παρουσιάστηκε, αυτή η συμφωνία μας παρουσιάστηκε σαν η λύση ε, για την κρίση. Ότι θα θα δώσει ωφέλη, θέσεις απασχόλησης, όταν οι μελέτες αντικτύπου που πραγματοποιήθηκαν στην καλύτερη υπόθεση δείχνουν ότι είναι πολύ μικρή αύξηση του ΑΕΠ. Μιλάμε για 545 ευρώ σε κατά οικογένεια το χρόνο, μεγαλύτερα έσοδα, έναντι τίνος τιμήματος, δηλαδή εναρμονίσεως όσον αφορά τους κανονισμούς μας και την νομοθεσία μας που προφανώς ξεκινώντας από διαφορετικούς κόσμους όπως είναι ο ευρωπαϊκός κόσμος βασίζεται στην αρχή της πρόληψης και το αμερικανικού κόσμο, όπου το βάρος απόδειξης βρίσκεται στην αγορά και στον καταναλωτή και στην εταιρεία που θα πρέπει να αποδείξει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν η χημική ουσία είναι επιζήμιο για την υγεία είναι εντελώ διαφορετικοί κόσμοι τόσο μακριά που με δυσκολία προσπαθώ να καταλάβω ε, ποια είναι τα πεδία εναρμονίσεως και ταύτισης μπορούμε να βρούμε. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και ελάχιστα γνωρίζουμε διότι δεν ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, πολύ συχνά παρουσιάζεται μόνο αποκλειστικά ευρωπαϊκή θέση, που βέβαια σίγουρα έχει μια οπτική γωνία προστασίας, ε, τα, τις και τα επίπεδα προστασίας που ήδη έχουμε, που είναι αρκετά υψηλά. Και ανοίγω και μια παρέθεση, όπως είπε η κυρία Ριβαζή, και η ΕΦΣΑ ίδια έχει πολλές, περιέχει πολλές σκιές και δεν πρέπει να, ε, δεν πρέπει να αυτό και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να παίξει θεμελιώδη ρόλο όσον αφορά τις επραγματεύσεις όμως δεν ελήφθη υπόψη επαρκώς μέχρι τώρα. Η Γενική Διεύθυνση Trade ε, οργάνωσε 129 συναντήσεις με τα λόμπι και τις πολυεθνικές και κλεισμένο των θυρών και ελάχιστα συναντήθηκε με τις, εκπροσώπησεις, με τις εκπροσώπους των πολιτών και της ΜΚΟ. Και η ίδια αναγνώριση, ε, την ίδια ανησυχία εξέφρασε και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής που είπε ότι το επίπεδο πρόσβασης στις πληροφορίες ποικίλει ανάλογα με τους συνομιλητές και με τους φορείς συμφερόντα με άλλα λόγια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τέλος, και εγώ λέω η ρήτρα του ISDS είναι κάτι πολύ επικίνδυνο που υπονομεύει την κυριαρχία των κρατών μελών. Είναι ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να μείνει εκτός της συνθήκης. Ε, διαφορετικά θα είναι εντελώς ε, εσφαλμένο. Ευχαριστώ Λεωνόρα. Σολεδάδο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εξ ονόματος ε, του συναδέλφου που είναι στο Παναμά. Ο συνάδελφος Ζουντιτ ε, είχε αναλάβει να παρουσιάσει τη θέση μας. Αρχικά, αλλά τον αντικαθιστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαλέσα. για την έκθεση που παρουσίασε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα για την παρουσία του. διότι εκφράζει τις ανησυχίες και άλλων πολιτών. Θα ήθελα να αναφερθώ στα πλέον σημαντικά κατεμέ ζητήματα. Ο στόχος της TTIP είναι να τονωθεί το εμπόριο και οι επενδύσεις και εμπορικέ σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ της Αμερικής. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο ένας από τους στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ε, προστατεύσει το υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Να προστατεύσει και να κατοχυρώσει τα υψηλά πρότυπα που ισχύουν σε πολλούς τομείς της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επίσης το ειδικό βάρος που έχουν εταίροι όπως η Κίνα, πέρα από τις ΕΠΑ. Ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να συνάψουμε μια συμφωνία με έναν μεγάλο εταίρο όπως ε, η ΕΠΑ. Δεν θέλουμε όμως σε πάση θυσία να υπογράψουμε μια συμφωνία εάν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα πρότυπα, τους κανόνες που έχουμε στον τομέα του περιβάλλοντος, ε, της προστασίας των καταναλωτών, της εσωτερικής αγοράς, της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, των προσώπων. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να τεθεί εν κινδύνο η πολιτιστική ποικιλομορφία, τα, οι δημόσιες υπηρεσίες. Ε, αυτά είναι κόκκινες γραμμές για μας και πρόκειται να εμείνουμε στη θέση μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το θέμα της διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Βάσει συνθήκη της Λισαβόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα για να διαπραγματεύεται και να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες. Η θέση σε ισχύ της ε, συμφωνίας, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, θα επέλθει μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Προβλέπεται δηλαδή έλεγχος κοινοβουλευτικός και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαφυλάξουμε τη διαφάνεια και τα πρότυπά μας. Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων έγινε το 2013 ακολούθησαν 8 γύροι διαπραγματεύσεων και έπονται και πολύ περισσότεροι. Μετά από κάθε διαπραγματευτικό γύρο ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα εκδώσουμε και ένα ψήφισμα για το σημείο στο οποίο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις για την TTIP. Δεν ισχυρίζομαι ότι επικρατεί απόλυτη διαφάνεια στην ε, διαδικασία διαπραγματεύσεων. Όμως, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτούς που ισχυρίζονται ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Υπήρξε μια καθυστέρηση και δεν δημοσιεύθηκε άμεσα το, η διαπραγματευτική εντολή. Αυτό είχε ένα αντικό αντίκτυπο στην αρχή της, διαδικασίας, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες είναι δυνατή πλέον για όλα τα μέλη, όχι μόνο της Επιτροπής Αναφορών, και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ίντα, με πρόκειται αποκλειστικό προνόμιο των συντονιστών. Θα πρέπει να επιδιώξουμε τα ίδια πρότυπα διαφάνειας και για τις υπόλοιπες εμπορικές συμφωνίες. Να θυμίσω ότι υπάρχει και μια ομάδα εργασίας στα πλαίσια της Επιτροπής ΙΝΤΑ για τη διαφάνεια. Η διαφάνεια και το θέμα της ε, διαιτησίας είναι ζητήματα που απασχολούν ιδιαιτέρως ε, την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Έχουμε ήδη 150.000 υπογραφές κατά του νέου ε, μηχανισμού διαιτησίας για τις διαφορές επενδυτού κράτους υπάρχει κινητοποίηση και νομίζω ότι η εθνική κυριαρχία και οι ένομες τάξεις των κρατών μελών θα μπορέσουν να παραμείνουν σε ισχύ ούτως ώστε να προστατευτούν οι επενδυτές μας ε, στη ΣΥΠΑ. Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι μάλλον ευίωνες. Να ευχαριστήσω κλείνοντας τον κύριο Βαλσάν για το σχέδιο έκθεσης, να ευχαριστήσω τον αναφέροντα για την παρουσία του στη σημερινή συνεδρίαση και ελπίζουμε όλοι ότι η νέα συμφωνία θα ε, ε, τηρεί πλήρω ε, τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωση σε όλους τους τομείς. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία που αναφέρθηκαν και ίσως ο συνάδελφος θέλει να αναφερθεί συγκεκριμένα στα τρόφιμα και την ασφάλεια τροφίμων. Πρώτον, το είπα και πριν, δεν συμβαίνουν εν κενό αυτές οι διαπραγματεύσεις. Θέλω να το τονίσω αυτό. Η εντολή είναι σαφή στο τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν, σαφή τα πράγματα και ο στόχος επίσης ε, και όσον αφορά και τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και τη στρατηγική αξία. Δεν θα τα επαναλάβω όλα αυτά. Δεύτερον, δημοκρατικός έλεγχος. Πρέπει να είμαστε σαφείς τι λέμε εδώ πέρα. Έχουμε μία έντολη, διαπραγματευόμαστε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις ξεκινάει η διαδικασία κύρωσης και εκεί πέρα έχουν πλήρεις αρμοδιότητες ε, τα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Οπότε εσείς και οι συνάδελφοί σας έχετε τον τελευταίο λόγο. Είναι σαφές. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι εννοείται ότι δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και δεν περιμένουμε την τελευταία στιγμή βεβαίως. Υπάρχει ο ρόλος των συναδέλφων σας στην Επιτροπή Ίντερ. Νομίζω υπήρχε και η Επιτροπή Παρακολούθησης ε, που συστάθηκε εκεί πέρα, η οποία παρακολουθεί αυτές τις διαπραγματεύσεις λεπτομερέστατα, με πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Υπάρχουν ε, απενημερώσεις, προενημερώσεις, ε, οπότε νομίζω πως ο δημοκρατικός έλεγχος υπάρχει και οπωσδήποτε εσείς και οι συνάδελφοί σας έχετε τον τελευταίο λόγο. Ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω το θέμα της εντολής γιατί λέτε πως η Κομισιόν δεν δημοσίευσε την εντολή. Η εντολή είναι ένα έγγραφο του Συμβουλίου που παραδίδεται στα κρατη Εμείς ζητάμε τη δημοσίευση της εντολής. Το Συμβούλιο δεν ήθελε. Η τελική απόφαση είναι του Συμβουλίου και αυτό την έλαβε όπως έχει κάνει και σε άλλες διαπραγματεύσεις ε, παραδείγματο χάρη στι διαπραγματεύσει τη ΤΙΖΑ, τι λεγόμενε. Η κυρία Οράιλι, η συνήγορος του πολίτη, είπε πως είναι ικανοποιητικό το επίπεδο ε, διαφάνειας και είπε επίσης πως ε, χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο επίπεδο ε, απορρίτου εμπιστευτικότητας. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ε, η σωστή ισορροπία μεταξύ δημοσιότητας, δημοσιοποίησης των κειμένων στο μέτρο του δυνατού, αλλά βεβαίως διατηρώντας την απαραίτητη εμπιστευτικότητα για να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία η οποία θα είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, απορρίπτω το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προνομιακή ε, μεταχείριση. Νομίζω πως όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν και από την τυζή της ΑΝΚΟ. Κάθε ομάδα, πολίτης, ένωση, ΜΚΟ, επιχειρηματίες έχουν την ίδια πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τελευταίο, επειδή αναφέρθηκε, δεν θέλω τώρα να μπω στις λεπτομέρειες του ISDS και της προστασίας των επενδυτών, γιατί υπάρχει μια συζήτηση αύριο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα. Απλά θα ήθελα να πω πως η διαβούλευση που έγινε είναι η βάση για τη μελλοντική δουλειά μας. Κοιτάξαμε όλες τις απαντήσεις που λάβαμε, 149.000 δεν απορρίψαμε καμία, δεν είπαμε πως κάποιες δεν μετράνε γιατί ήταν ε, διπλές, ε, τις κοιτάξαμε όλες, βγάλαμε τις ιδέες, τις προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει, τις προτάσεις για βελτίωση. Ε, καταλήξαμε σε τέσσερις τομείς και αυτοί οι τέσσερις τομείς και άλλοι τώρα θα συζητηθούν με τους συναδέλφους σας στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και στα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε σε μια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις αυτές. Αυτά νομίζω ο συνάδελφος από την DG Σάνκο θα ήθελε να πει κάτι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα να αναφερθώ σε κάποια από τα ζητήματα που είπε ο συνάδελφος ε, και το κοινό. Η αρχή της προφύλαξης. Όπως είπαμε δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε την θέση μας. Είναι στο κείμενό μας και παρά το ότι οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν ε, δεν την αναγνωρίζουν, την εφαρμόζουν αυτή την αρχή για τις εξαγωγές μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το χαμόν σεράνο, το προσούτο, ε, όλα αυτά τα... Αλλαντικά αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα γιατί ακριβώς εφαρμόζουν ε, οι ΙΠΑ τις αρχές ε, της προφύλαξης όσον αφορά τα αλλαντικά αέρος. Οπότε ούτε η ΕΠΑ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουν την προσέγγιση τους για την αρχή της προφύλαξης. Νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, που μπορούμε να δούμε ακριβώς για να συντονίσουμε την συμπεριφορά μας στο πλαίσιο του ρυθμιστικού μας περιβάλλοντος και αν λάβετε υπόψη τους τρεις τομείς όπου είναι πιο σαφές ε, το αμερικανικό ενδιαφέρον, δηλαδή ορμόνες, αντιμικροβιακή θεραπεία και την ε, ακτινοβόληση, πράγματι εκεί πέρα θα ε, προστατεύσουμε τους καταναλωτές μας. Τώρα, αντιμικροβιακή μεταχείριση, η οποία γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης ε, νομίζω μπορεί να είναι υποφελής. Ε, αν δούμε ένα από τα ζητήματα, παραδείγματο χάρη, το οποίο απασχολεί πολύ το κοινό, το τι γίνεται με τα πουλερικά. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εάν δείτε τα δεδομένα για τα κάμπυλοβακτήρια που παρουσιάζει η Αρχή Προστασίας Τροφίμων, έχουμε 200.000 περιπτώσεις κάθε έτος ε, κάμπυλοβακτήριασης βεβαιωμένες περιπτώσεις. Επίσης η ΕΦΣΑ λέει πω υπολογίζονται οι περιπτώσεις ότι φτάνουν μέχρι και τα 9 εκατομμύρια κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προκαλούν πέρα από τα θύματα 1 έως 5 εκατομμύρια ευρώ κόστος στο σύστημα υγείας. Οπότε ε, είναι τέλειο το σύστημά μας από την πλευρά αυτή ή μήπως μπορούμε στο πλαίσιο αυτό με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ η οποία όπως ξέρετε βασίζεται σε ανεξάρτητους ειδικού. Ε, μήπως λοιπόν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συζήτηση για να βελτιώσουμε περαιτέρω το σύστημα ασφαλείας τροφίμων. Νομίζω πως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε. Επίσης, ε, ε, μιλήσατε για παραλληλισμούς μεταξύ ΙΠΑ, ε, Καναδά με συγχωρείτε και ΙΠΑ. Δεν χρειάζεται λοιπόν ανησυχία γιατί το ό,τι κάναμε με τον Καναδά κάνουμε και με τις ΙΠΑ. Η συμφωνία αυτή η TTIP δεν είναι η πρώτη συμφωνία με τις ΙΠΑ στον τομέα ασφάλειας τροφίμων, έχουμε μια κτηνιατρική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, όπως έχουμε και με τον Καναδά, που ισχύει από το 1999. Οπότε συνεργαζόμαστε με τη ΣΥΠΑ με τρόπο δομημένο εδώ και 15 χρόνια. Αυτό το οποίο κάναμε με τον Καναδά είναι αυτό το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε με τις ΣΥΠΑ. Δηλαδή να πάρουμε αυτή την κτηνιατρική συμφωνία που ε, είναι η βάση των σχέσεών μας και να την μεταφέρουμε στα ε, υγειονομικά και φυτογειονομικά κεφάλαια της συμφωνίας ΣΕΤΑ με τον Καναδά και ΤΙΤΙΠ με τις ίπα. Τι είναι λοιπόν το υγειονομικό κεφάλαιο, ένα κτηνιατρικό και ένα φυτογειονομικό κεφάλαιο. Πρέπει λοιπόν να κοιτάμε περισσότερο τις ευκαιρίες. Ε, οι κίνδυνοι περιορίζονται, αλλά οι ευκαιρίες είναι τεράστιες. Ε, ήδη σήμερα είπα με TTIP ή χωρίς μπορούν να εξάγουν όλα τα προϊόντα ζωικής ή φυτικής προέλευσης επειδή το σύστημά μας είναι το πιο ανοιχτό παγκοσμίω. Ανεξαρτήτως του αν υπάρχει ειδημερή συμφωνία, αν δούμε τα ίδια προϊόντα που μπορούμε εμείς να εξάγουμε στη ΣΥΠΑ, δεν μπορούμε να εξάγουμε παραδείγματος χάρη προϊόντα αυγών Επίσης ε, δεν μπορούμε να εξάγουμε προϊόντα με παστεριωμένο γάλα, βοδινό και πρόβιο Και για λαχανικά χρειάζεται και κάθε κράτος μέλος να περάσει μια δικασία 10-15 ετών για να κάνει εξαγωγή ε, ένα κράτος μέλος μήλα. Αυτό το οποίο θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε είναι περισσότερες ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα στο σύνολό της και όχι για τα κράτη-μέλη τα οποία σήμερα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο για να κάνουν μια εξαγωγή στη ΣΥΠΑ. Υπάρχει και μια συμφωνία ελευθέρου μπορείου μεταξύ δύο μπλοκ. Και αυτό είναι, αυτή είναι η λογική. Κάνετε εξαγωγέ, κάνουμε και εμείς εξαγωγές, σεβόμενοι ο καθένας τους κανόνες του άλλου. Οπότε, οι κίνδυνοι είναι πολύ περιορισμένη, όπως σας είπα, ε, η απόδειξη ε, είναι σαφής, έχετε τα 15 χρόνια δομημένων σχέσεων στον κτηνιατρικό τομέα με ΙΠΑ, με Καναδά, με Νέα Ζηλανδία. Αυτό κάνουμε γιατί αυτό είναι το αριθμιστικό μας πλαίσιο. Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εκτός του ρυθμιστικού μας πλαισίου. Ακόμα και στο πλαίσιο, όπως είπαμε, διμερών εμπορικών σχέσεων. Ευχαριστούμε την Κομισιόν. Yeah. Από τους βουλευτές δεν θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. Τον λόγο έχει λοιπόν ο αναφέρον για δύο λεπτάκια. Μάλιστα, να απαντήσω σύντομα σε αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν. Είναι νομίζω συμπτωματικό της όλης κατάστασης, ενδεικτικό της όλης κατάστασης ε, ε, το χάσμα αυτό μεταξύ εκπροσώπων και πολιτών. Και βλέπετε ακριβώς το πώς ήρθε η TTIP ε, στο προσκήνιο. Κρύψατε τα πράγματα όσο το δυνατόν περισσότερο και μετά είχαμε μια εκστρατεία διαφημιστική. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε τώρα να μας πείτε ότι υπάρχει διαφάνεια και αναφέρθηκε ήδη, ε, αναφέρθηκε δηλαδή κάποιες αίθουσες ανάγνωσης στους οποίες δεν επιτρέπεται τα αντίγραφα. Μα τι διαφάνεια είναι αυτή. Ή λέτε πως δόθηκε μία έντολη και ο περισσότερος κόσμος τότε δεν ήξερε ότι υπάρχει τέτοια συμφωνία. Προσπαθήσατε δε να πείτε πως η δικιά μου η αναφορά αφορά μόνο την προστασία των τροφίμων και των καταναλωτών. Και όμως είναι πάρα πολύ περισσότερα τα πράγματα. Το θέμα είναι όπως είπα συντάξεις, υγεία, εκπαίδευση. Αν δούμε όμως πως ε, έχουμε τομείς που πάνε για εναρμόνιση που δεν επιτρέπεται να εναρμονίζονται ακόμα και τα πνευματικά δικαιώματα στη ΣΥΠΑ επιτρέπεται η πώληση των πνευματικών δικαιωμάτων ενώ στην Ευρώπη είναι πάντα με τον δημιουργό. Πρέπει να σας πω πως ε, είχα πάει και στις ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον και είδα εκεί πέρα τι προσπαθούν να κάνουν παρά το ότι είναι πάρα πολύ ε, πιο διαφανής η διαδικασία. Αν δούμε τώρα τη συμφωνία με την Νότια Κορέα δείτε εκεί πέρα το τι αναφέρεται για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τελείως πουλημένο, τελείως ε, ξεπουλάτε την ιδιωτική σφαίρα του πολίτη. Όχι, πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τις διαμαρτυρίες του κόσμου. Μην απορείτε λοιπόν για το ότι κάθε μέρα όλο και περισσότερες ΜΚΟ είναι κατά της συμφωνίας αυτή αυτής όταν την ε, παρουσιάζεται ως μια συμφωνία της διαφάνειας και της συμμετοχής ενώ είναι κάθε άλλο από αυτό. Ευχαριστούμε. Κύριος ε, Βαλέσσα ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Κύριε Κράμερ, είστε βέβαιος ότι μεταξύ Ευρωπαϊκού Λαού και Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το Ευρωκοινοβούλιο και από εμά εξαρτάται να αποφασίσουμε αν θα δεχτούμε το τι τύπη θα το απορρίψουμε. Στο τέλος λοιπόν, το δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξασφαλίσει το ότι δεν θα συμφωνήσει επί μια συμφωνίας που δεν θα είναι υποφελής για τους λαούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη πρόταση, την εξής. Σας προτείνω να στείλετε στον αναφέροντα μετά την ψηφοφορία της Δευτέρας την, ε, ε, ε, μετά την ψηφοφορία του κειμένου στην Ίντα. Θα στείλουμε το κείμενο στον αναφέροντα και η ψηφοφορία για την Επιτροπή Αναφορών 23 Μαρτίου, η προθεσμία για τις τροπολογίες, ψηφοφορία 16 Απριλίου και ψηφοφορία στην Ίντα το μήνα Μάιο. Ιδού λοιπόν το χρονοδιάγραμμα για την Επιτροπή των Αναφορών. 23 Μαρτίου για τις τροπολογίες στην Επιτροπή Αναφορών 16 του Απριλίου στην Επιτροπή Αναφορών Ψηφοφορία και μετά την Επιτροπή στην Επιτροπή Αναφορών θα στείλουμε στους αναφέροντες όλη, όλη τη, όλα τα έγγραφα η την αναφορά και της, ε, της δικής μας Επιτροπής και της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ ώστε να μπορούν να έχουν τις πληροφορίες μετά την έγκριση της εκθέσεως και έτσι τελικά θα κλείσει η αναφορά. Πολύ καλά λοιπόν. Θα τα πούμε ξανά στις 3 ακριβώς. Παρακαλώ να είστε ακριβείς για να μπορέσουμε περισσότερο χρόνο για τις αναφορές. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.